Voilà, Καλησπέρα σας. Ξεκινάμε. Τα χθεσινά πρακτικά και τα ε, εγκεκριμένα κείμενα έχουν μοιραστεί. Υπάρχουν παρατηρήσει, Όχι. Οπότε θεωρούνται ω εγκεκριμένα τα πρακτικά.